Je vous σιγά σιγά και ετοιμάστε τις κάρτες σας για ψηφοφορία διότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς κάρτα.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 έχουμε διάφορες προσωπικότητες της Επιτροπής μας. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μίτσελ και την κυρία Εύα Ζολή που είναι υποψήφοι στις ε, χώρες τους αντιστοίχως. Και θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τις κάρτες σας για να κάνουμε μια δοκιμή. Η κυρία Τζίμερ. Θέλω παρακαλώ να ζητήσω πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία να μπορέσω να κάνω κάποια παρατήρηση επί της ψηφοφορίας. Ωραία. Μπορείτε να το πράξετε τώρα, προτού ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τη στήριξη στην ε, επεξεργασία αυτής ε, της εκθέσεως και επιτύχαμε καλούς συμβιβαστικούς, καλές συμβαστικές προτάσεις και τροπολογίες και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα με τους γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς αλλά όσον αφορά την τροπολογία 66 ε, προσπαθήσαμε να τη συμπεριλάβουμε, αλλά ε, ποτέ δεν αντέδρασε και το επισημένο, διότι ε, αν υπερψηφίσει κανείς την τροπολογία 66, αυτό θα αμφισβητήσει την ε, ε, ε, την συμβιβαστική μας τροπολογία age ήταν. Οπότε θα παρακαλούσα να συμφωνήσουμε και να έχετε υπόψη σας ότι αν υπερψηφιστεί η τροπολογία 66 θα αμφισβητηθεί η συμβιβαστική μας τροπολογία. Λοιπόν, ε, ας ελέγξουμε τώρα την ε, λειτουργία των καρτών. Μπορείτε να ψηφίσετε δοκιμαστικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ακόμη ένα άτομο. Και άλλο ένα. Λοιπόν, λίγη ψηφοφορία. θα προχωρήσουμε πιο αργά γιατί έχουμε πολλές συμβιβαστικές. Ο κύριος Μπέρμαν καταρχήν. Θα ε, ψηφίζουμε κύριε Μπέρμαν, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ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 δεν έχουμε τα ίδια χαρτιά. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ε, ομαδικά μέχρι το 16 υπέρ κατά αποχές όλα με την συμβιβαστική Β όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται και φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική Γ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι όμως βέβαιη, ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Ξεκινάει. Λίγοι. Υπέρ. Παρακαλώ μπορείτε να μου στείλετε ένα τεχνικό. Θα αλλάξω κάθισμα κυρία Πρόεδρε λέει ο κύριος Νιούτον Τζον τον ε, μπορούμε να προσθέσουμε την ψήφο σας. Ήσασταν υπέρ ή κατά. Δεν αλλάζει τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τροπολογία 21 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 22 απεσύρθη. Είμαστε τώρα στη συμβαστική D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Καταπίπτει. 25. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 25. Λίγοι. 12 υπέρ, 11 κατά, εφόσον ο κύριος Νιούτον Ντάν είναι αντίθετος. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, καταπίπτει καταπίπτει η συμβιβαστική ε εφόσον υπερψηφίστηκε η τροπολογία 26 και φτάνουμε στην 30. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίθηκε 26 η συμβιβαστική ε καταπίπτει και άρα ούτε η 27, 28 και 29 δεν ε, καταπίπτουν εφόσον δεν υιοθετήθηκε η συμβιβαστική ε. Άρα οι τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονταν σε αυτή τη συμβιβαστική δεν ε, καλύπτονται. Ναι, αλλά λέει ότι καταπίπτουν εάν η τροπολογία 26 ε, άρα η 26 δεν ε, εφαρμόζεται μόνο εις ε, τη συμβιβαστική ε αλλά και σε όλες τις άλλες. Ναι, όντως ε, δεν εμφανίζεται ευκρινώς εις το φύλλο της ψηφοφορίας. Ψηφίσαμε λοιπόν τώρα την 30. 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Λοιπόν, 36 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά δεν είμαι βεβαία ηλεκτρονικός έλεγχος για την 37. Λίγη ψηφοφορία. Κύριε Νιούτον Ντάν, ψηφίσατε. Μάλιστα. Είσαστε υπέρ. 12-11, άρα ε, εγκρίνεται. Η κυρία Τσίμερ ζητάει το λόγο. Λοιπόν, Έκανε ένα λάθος, ήθελα να υπερψηφίσω, οπότε εγκρίνεται σαφώς. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, 38 υπέρ, κατά, ελέγχουμε γιατί δεν είναι ακριβό, δεν είναι σαφές. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38, λίγη, απερίφθη. 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ε, ε, τροπολογία 3 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Επιτροπή Γεωργία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο σχετικά με την τροπολογία 1 της Επιτροπής Γεωργίας ε, ξεκινά, λίγη, ενεκρίθη. Συμβασική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε έρχομαι στη 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ είναι ταυτόσημα με τον 42. Άρα εγκρίνεται. 44 υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια για να μπορούμε να μετρήσουμε σωστά. Κατά. Δεν σηκώνει κανείς το χέρι του, νομίζω ότι απερίφθη, αλλά θα ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Ενεκρίθη. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Γεωργία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είμαστε στην συμβιβαστική age. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτα. Και ερχόμαστε στην 61 υπέρ. Κατά. Για να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο σχετικά με την 61. Ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη. Κύριε Κάσμαν, δεν λειτουργεί το μηχανάκι σας. Απερίπτεται ούτως ή αλέως. Πού ήμασταν λοιπόν, ε, μάλλον 12-12, άρα απορρίπτεται. Ούτε εκεί λειτουργεί. Την έχετε βάλει ανάποδα κύριε Κάσουμαν την κάρτα σας ψηφοφορίας. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στην 65. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω ότι ενεκρίθη, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 65. Λίγοι. συμφωνήσατε, ε, είσαι στόμος αντίθετος. Οπότε είναι 11 υπέρ, 13 κατά, απορρίπτεται. Παρακαλώ όμως να δοκιμάσετε την κάρτα σας για του κυρίου Μπέρμαν αλλάζοντας ε, ο κύριος, ε, ο τεχνικός ε, πήρε την κάρτα μου για να την ελέγξει και δεν έχω κάρτα αυτή τη στιγμή. 66 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είμαι όμως βέβαιη. Τροπολογία 68, ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη. Απερι... Εσείς υπερψηφίσατε απερίφθη παρόλα αυτά, γιατί είμαστε ε, ισοψηφία. Ε, 69 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχο με συγχωρείστε, αλλά όταν υπάρχει μία ψήφος διαφορά πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά για την τροπολογία 69, λίγη. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά η δικιά μου κάρτα δεν δουλεύει. Εγώ καταψηφίζω όλα αυτά απορρίπτεται. Τώρα ότι η δικιά μου κάρτα λειτουργεί. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 ε, υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 71 ξεκινά. Τώρα όμως λειτουργεί. Λίγη ψηφοφορία. Εσείς υπερψηφίζετε. Απερίφθη. Γεωργία 19 υπέρ κατά αποχές 13 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε να ψηφίσουμε συνολικά τις ε, τροπολογίες 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γεωργία 18 υπέρ ε, της Γεωργίας όλες δηλαδή 18 μέχρι 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, τροπολογία 83 ξεκινά η ψηφοφορία λίγη εγκρίνεται. 18 υπέρ, 6 κατά. 84 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Γεωργία 5 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 85, μάλλον η 85 αποσύρεται είναι δικιά μου και απεσύρθη. Συμβιβαστική J, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τώρα είμαστε στην ε, τροπολογία Γεωργίας 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 93 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, ξεκινά η ψηφοφορία, λίγη. Απερίφθη. Απερίφθη παρόλα αυτά. Ε, Γεωργία 9 ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...96, τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έχουμε μία προφορική τροπολογία εδώ και δίνω το λόγο στον κύριο Σβένσον. Κύριε Σβένσον έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η προφορική τροποποίηση έχει ως εξής. εκφράσει την ανησυχία της ότι το 2008 η χρονιά της κρίσης ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη παραγωγή στην ιστορία του κόσμου. Ε, αυτό δείχνει τον αρνητικό ρόλο της κερδοσκοπίας ε, στους δείκτες τιμών των αγαθών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το 100 καταπίπτει και περνάμε στην 101α, υπέρ, κατά, απορρίπτεται 102, κατά, εγκρίνεται 103, υπέρ, κατά, αποχή, θα ελέγξουμε Ανοίγει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αγκρί 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχή. Αγκρίνεται 104. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 105 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 12 και 12. Απορρίπτεται συνεπώς. Τροπολογία 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά δεν γνωρίζω 111 ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει κλείνει ψηφοφορία 12 και 12 συνεπώς απορρίπτεται τροπολογία 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αγκρί 7, γεργή 7 υπέρ, κατά, οι αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική L, λάμδα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 120 τροπολογία υπέρ κατά. Εγκρίθηκε 121 υπέρ κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ξεκινάει. Έχει κλείσει για, το, για την 121. 12 και 12. Συνεπώς απορρίπτεται. Αγκρί 10, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αγκρί 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά. Ε, σηκώστε καλά τα χέρια. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 122 ξεκινάει. Λίγη ψηφοφορία. 11 και 12 απορρίπτεται. Συμβιβαστική M. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται 123 τροπολογία, ε, συγγνώμη, 127 τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, ελέγχουμε, ε, ανοίγει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, 12 και 12, απορρίπτεται. Τροπολογία 128 υπέρ, κατά. Ε, θα ελέγξουμε, ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη η ψηφοφορία. 11 και 12 απορρίπτεται. Μέχρι και... Λοιπόν, μαζικά μέχρι την 133 και την 133 υπέρ. Θα το κάνουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, από την 129 μέχρι την 133 ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 12 και 12 απορρίπτονται. 134 τροπολογία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά. Δεύτερο μέρος ελέγχουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Συνεπώς 12-11 εγκρίνεται. Τρο... Παράγραφος 19. Υπέρ κατά... Ε, ε, λοιπόν, συγγνώμη, τροπολογία 135. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική, ε, ξεκινάει, λίγη ψηφοφορία, 12 και 12 απορρίπτεται, τροπολογία 130, 140, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε Σηκώστε καλά τα χέρια γιατί έτσι όπως γίνεται δεν ξέρουμε αν είστε υπέρ κατά 140 ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 140. Με Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κυρία Ζήμερ, θέλατε το λόγο. Ναι. Εδώ επανέρχομαι διότι μία τροπολογία δεν έχει ψηφιστεί 137. Από την 136 πήγαμε κατευθείαν στην 138. Με συγχωρείτε. Οπότε τώρα ψηφίζουμε την 137. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα έχω χαθεί λιγάκι. Βρισκόμαστε στην 142 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε, ανοίγει ψηφοφορία για την 142, κλείνει, 13 απορρίπτεται τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά ελέγχουμε ξεκινάει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία ναι και 15 απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει Λίγη ψηφοφορία. 12 και 12 απορρίπτεται. Αγκρί 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. 150 ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει. Κλείνει. 8 και 16 απορρίπτεται. Τροπολογία 151, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ελέγχουμε, 151 ξεκινάει. Η ψηφοφορία, κλείνει η ψηφοφορία. 14-10 εγκρίνεται, 152 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, 153 υπέρ, κατά. Αποχές ελέγχουμε, 153 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 10 και 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 154. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 155 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται, 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία 12 και 12 απορρίπτεται τροπολογία 159 σε δύο μέρη για το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά Ελέγχουμε το δεύτερο μέρος, ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το δεύτερο μέρος του 159, κλείνει η ψηφοφορία, 12 και 12 απορρίπτεται. Γεωργία 2, εγκρί 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, εγκρί 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 160 τροπολογία υπέρ, κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά Νομίζω ότι είναι υπέρ 160 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 10 και 14 απορρίπτεται. Παράγραφος 15. Συμβιβαστική ομικρόν. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 161. Περνάμε στην τροπολογία 163. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αγκρι 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική π ποιος είναι υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται τροπολογία 166 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία 12 και 12 συνεπώς απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία για την 168, 12 και 12 συνεπώς απορρίπτεται. Τροπολογία 169 υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 14 και 10 εγκρίνεται. Τροπολογία 170 υπέρ, κατά. Α, ε, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 13 και 12 εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η τελική ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 18 και 6 συνεπώς εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη ε, κυρία Τσίμερ.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 Je vais continuer avant que tout le monde s'échappe. Συνεχίζω, μην φεύγετε όλοι. Σας παρακαλώ, ε, αφήστε όσους ε, εργάζονται να εργαστούν και φύγετε από την αίθουσα εάν δεν θέλετε να μείνετε, το οποίο δεν το συστήνω. Η πολιτική της άδεια καρέκλας δεν είναι καλή. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας έχει αποφασίσει να συντάξει μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για το τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου. Παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο να μην μιλάτε. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας έχει αποφασίσει να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας για το τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου για την αντιμετώπιση της, ε, στο φόρουμ του Νοεμβρίου στο Πουσάν θα μας παρουσιάσει σήμερα τις κύριες ιδέες ε, της εκθέσης του ε, συναδελφό μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του και για, έναν, για την παρουσία ενός εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών, κυρία Κρό, διευθύντρια της ΜΚΑΠΟΑ Πλαν έρόπ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που τώρα ξεκινάει να συζητιέται στο Συμβούλιο δεν έχει ακόμα κληθεί να εκφράσει την άποψή του. Θα δώσω λοιπόν το ε, λόγο στον κύριο Πρέντα, στον εισηγητή. Ε, προσπαθήστε παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τρία σημεία όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης που σας παρουσιάζω σήμερα. Πριν από ένα μήνα το είχαμε συζητήσει σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να εξετάσουμε ε, που εντάσσεται στη συζήτησή μας. Ε, όπως γνωρίζετε σήμερα απέχουμε τέσσερις μήνες από το φόρουμ του Πουσάν και με την προοπτική της προετοιμασίας αυτής της συνεδρίασης θα ήθελα να επισημάνω δύο σημαντικές εξελίξεις ε, οι οποίες έλαβαν χώρα μετά την τελευταία μας συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα, ο, ο ΣΑ είδε τα πρώτα αποτελέσματα. Δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απομένουν πολλά να γίνουν για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Αυτές οι δεσμεύσεις ε, είναι σημαντικές και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της αρρωγής και τη διαφάνεια των εταιρικών σχέσεων που ασχολείται με όλο και με σημαντικότερες ποσότητες ε, έργου. Παγκοσμίως, οι βελτιώσεις που έχει φέρει η δήλωση των Παρισίων δεν έχουν βοηθήσει στην βελτίωση του φόρτου διαχείρισης της αρρωγής, όπως ελπίζαμε στις 22 Ιουνίου η πρώτη έκδοση του τελικού εγγράφου για το τέταρτο φόρουμ ε, δημοσιεύτηκε από την Ομάδα Εργασίας για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας. Την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους στον ΩΣΑ. Ε, δείχνει το έγγραφο αυτό μια αλλαγή των διακυβευμάτων και των θέλοντας ε, να εμβαθύνουμε τις δεσμεύσεις του Παρισιού αναδεικνύει την ανάγκη για μια, ένα νέο υπόδειγμα και μια νέα εταιρική σχέση. Επικεντρώνεται σε δεσμεύσεις όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης, και τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα της αρρωγής. Αυτή η πρώτη έκδοση του τελικού εγγράφου έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ακόμα για τα οποία πρέπει να γίνουν επιλογές από τους συμμετέχοντες στο φόρουμ στα τέλη Νοεμβρίου. Όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της αρρωγής, το δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης που έχω εκπονήσει και που έχετε στους φακέλους σας. Το πρώτο που θέλω να πω όσον αφορά το περιεχόμενο είναι ότι απαιτεί μεγάλη δέσμευση και συμμετοχή υψηλού επίπεδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Φόρουμ του Μπουσάν δεδομένων των διακυβευμάτων ε, της αποτελεσματικότητας της ε, βοήθειας ε, για τους επίτευξη των στόχων του 2015 είναι σημαντικό. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή στο Μπουσάν. Επίσης θα χρειαστεί η υλοποίηση άμεση των δεσμεύσεων του Παρισιού που εξαρτάται από την πολιτική βούλαση και από τη γραφειοκρατία. Χρειάζεται βούληση και διαφάνεια της αρρωγής. Επισημαίνεται επίση η δημοκρατική ανάληψη ευθύνη της αρρωγής και ο, να υπάρχει ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην παροχή της βοήθειας αυτής. Τρίτο σημείο, χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός στις χώρες αποδέκτες μεταξύ των εθνικών και τοπικών διαδικασιών ανάπτυξης και στο επίπεδο των παρόχων της βοηθείας. Το τελευταίο σημείο αφορά την ανάγκη βελτίωσης της, του καταμερισμού εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της απουσίας πολιτικής βούλησης. Έχουμε συζητήσει ήδη αυτό το ζήτημα του καταμερισμού των εργασιών. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία που χρειάζεται βάθυνση με τροπολογίε. Ε, ε, είμαι υποχρεωμένο να αναφερθώ σε αυτό, διότι η γραμματεία ήταν πολύ σκληρή και χρειάστηκε να διαγράψω ορισμένα σημεία. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, αποφάσισα να εμβαθύνω ορισμένα σημεία με τροπολογίε. στο 26 για παράδειγμα η αποτελεσματικότητα της βοήθειας για την ανάπτυξη ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την καινοτομία ε, άλλες πιθανές τροπολογίες ε, αφορούν το ζήτημα της ε, δημοσιονομικής στήριξης σε σχέση με τους αναδιόμενους παρόχους που ανέφερα την προηγούμενη φορά. Βελτίωση της διεθνούς κυβέρνησης σε περίπτωση διεθνούς εταιρικής σχέσης ε, ώστε, έτσι ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο κεκτημένο όσον αφορά την ε, παροχή της αρρωγής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάρλος για να ολοκληρώσω από τη Γραμματεία για την υποστήριξή του και αναμένω τα σχολιά σας, τις αντιδράσεις σας όσον αφορά τις τροπολογίες. Ε, ελπίζω να κάνουμε μια παραγωγική, μια επικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους για αυτό το ε, συναρπαστικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Σου. Σας θυμίζω ότι έχουμε καθυστερήσει σημαντικά. Δίνω την κυρία, το λόγο στην κυρία Σου για ε, πέντε λεπτά το πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ενίσταμε εναντίον αυτής ε, της ε, κατηγορίας. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ σήμερα το δίκτυο για την ε, ε, υγεία που ταρτίζεται από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ανά την Ευρώπη και ε, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να συνεργαστούμε. καλύτερη ενίσχυση το οποίο σημαίνει ότι ακολουθούμε αυτούς τους, αυτές τις αρχές και μετά είναι η, η ανοιχτή μέθοδος στα πλαίσια των αρχών των Παρισίων. Τώρα έχουμε Τώρα έχουμε τις αρχές της Κωνσταντινούπολης επίσης. και από το Μπουσάν τα μηνύματα είναι δημοκρατική ε, ιδιοκτησία και επίσης να αξιολογήσουμε αυτά τα κριτήρια. Να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και επαλήθευση. Αυτή η δημοκρατική ιδιοποίηση. θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όσον αφορά τις ε, δεσμεύσεις, την επαλήθευση και τη διαφάνεια. Επίσης, σε κρίση της ε, φτώχειας, Αυτό αφορά και την εποπτεία για αυτούς που εκτελούν τα προγράμματα. Ε, αυτό αφορά και τις μανάδες που τα παιδιά στις ε, κλινικές για εμβόλια. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει κάποια αρχιτεκτονική της δίκαιης ε, παροχής της βοήθειας, της ενίσχυσης. Η υγεία είναι τομέας όπου έχουμε κατευθύνει μεγάλο κομμάτι αυτής της βοήθειας. Προσπαθούμε εκεί να καλύψουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. Οι τρει τομεί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσά είναι πρώτα-πρώτα ο συντονισμό των δωρητών, εναρμόνιση, κατανομή εργασία στην Ένωση Θα πρέπει όμως να υλοποιούνται αυτά τα οποία εξαγγέλλονται. Για το... Ε, τα ποσοστά δεν αυξήθηκαν σε όσον αφορά την υγεία. και επίσης αυτή η κατανομή των ρόλων της εργασίας του έργου δεν θα πρέπει να καταλήγει στο να δίνεται στην υγεία μικρότερο κομμάτι αυτού του πόρου. Όσον αφορά αυτή τη δημοκρατική ιδιοποίηση επίση, έχουμε παραδείγματα για το κοινοβούλιο από την Ουγγάντα. Εκεί ε, ε, βγήκε μια δυναμική στρατηγική και η κοινωνία των πολιτών. Στο Σαλβαδόρ επίσης είναι ένα παράδειγμα πως έχουμε μια διαρθρωμένη διαδικασία και χρειάζεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, το κατάλληλο χώρο όπου να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών. Αλλά είναι και κατάλληλα διαδρομένα. Οπότε θα πρέπει οι πόροι στο Μαλάου, επίσης έχει αποδώσει αυτή η στρατηγική. Ε, όμως ε, η προοπτική value for money δεν στην Τανζανία ας πούμε όπου γίνονται εμβολιασμοί ανοσο, ανοσοποιητικοί εμβολιασμοί αλλά με πληρωμή. Να κλείσω με αυτό. Είναι τα δύο βασικά σημεία τα οποία θέλουμε να γίνουν προτεραιότητες για το κοινοβούλιο. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε μία διαρκή υποστήριξη όσον αφορά την ενίσχυση στον τομέα της υγείας, για την ευθυγράμμιση και για την ιδιοποίηση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πιάνουν τόπο αυτό το οποίο κάνουν στον κόσμο. Άρα θα πρέπει να τους αποθαρρύνουμε από το να αποσυρθούν τους δωρητές. Εμφανίζονται όλα αυτά βέβαια στο σχέδιο κειμένου, ε, θα πρέπει να επιμείνετε σε αυτές τις θέσεις και άρα θα πρέπει να δείξουμε στην κοινωνία ότι υπάρχει χώρος να υπάρχει αλληλεπίδραση για την ε, ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στους βουλευτές. Ξεκινάω από την κυρία Σνίνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ για το σχέδιο εκθέσεως, ευχαριστώ και την κυρία Σρό για τα σχόλιά της. Έχω δύο ανησυχίες. Ε, Καταρχήν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία παραπομπή σε ένα θέμα που θεωρώ αναγκαίο. Ο συνδυασμός του, της κλιματολογικής πολιτικής με την πολιτική ανάπτυξης. Θα υπάρχει κάποια παραπομπή στην κλιματολογική ε, πολιτική αλλά θα πρέπει να διατυπωθεί πιο σαφώς. Και δεύτερον πρέπει να αναφερθούμε σε στενότερη συνεργασία με το νέο περιβάλλον διότι η τελευταίος έχει ε, συντάξει πολλά έγγραφα σχετικά με αυτό το θέμα οπότε ενδέχεται να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον και είναι μια δυνατότητα την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση έχει τρία βασικά θέματα προσοχή, διαφάνεια και ακρίβεια και ο κύριος Πρέντα ανταποκρίνεται στις επιταγές αυτές. Πριν από τον Μπουσάν πρέπει να διατυπώσουμε σαφώς όπου θέλουμε να καταλήξουμε με την αναπτυξιακή μας πολιτική γιατί μαζί με τα κράτη-μέλη εμείς είμαστε διεθνώς ο μεγαλύτερος δωρητής και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην, στην αποτελεσματικότητα της βοήθειάς μας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπροσωπηθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτή τη διάσκεψη διότι πρέπει να έχουμε μετρήσιμους και ε, υπολογίσιμους στόχους οι οποίοι έχουν έναν μηχανισμό εφαρμογής, ε, ε, enforcement mechanism, ιδίως αν θέλουμε ε, να προχωρήσουμε και πέραν των στόχων του 2015. Θέλουμε να έχουμε δημοκρατικούς συμμετόχους οι οποίοι θα συμπράξουν, να συμπεριληφθούν τα εθνικά κοινοβούλια, η κοινωνία των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση διότι η βελτιωμένη περιφερειακή διαχείριση θα είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό που είπε η προλαλή ότι χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό με τους άλλους δωρητές και ιδιαίτερος με την Κίνα είναι πολύ σημαντικό αλλά αυτό προϋποθέτει ότι εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα υπάρχει μια καλύτερη, ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών διότι έτσι ε, θα μπορέσουμε να αναλάβουμε την ε, ευθύνη μας καλύτερα και τέλος θέλω να πω ότι εάν ε, θέλουμε να ελέγξουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη συμμετοχή. Ε, συζητήσαμε και τροπολογίες. Εγώ έχω μόνο μία τροπολογία να προσθέσω η οποία τονίζει την σημασία της διαφανείας στα πλαίσια της ε, International Aid Transparency Initiative Θέλω να ε, ευχαριστήσω την Global Health και τον εισηγητή. Το έγγραφό του είναι πολύ καλό για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στον Μπουσάν. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα συγχαρώ τον συγγραφέα της ε, εισήγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι στιγμής η όλη προσπάθεια χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα της βοήθειας, από μη κάλυψη των στόχων και από, και από αποτυχία στην στόχευση. Γι' αυτό νομίζω ότι η συμμετοχή στη διάσκεψη του Πουσάν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά δεν αποδεικνύει αυτόματα και την πολιτική βούληση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, την δικιά μας πολιτική βούληση. Γιατί πρέπει να υπάρχει και συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος τόσο από μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου, αλλά και από μέρους όλων των δωρητών. Διότι πολλά κονδύλια έχουν δοθεί μέχρι σήμερα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα τα οποία δεν χρησιμοποίησαν καθόλου προς όφελος των πληθυσμών τους. Παράλληλα πρέπει να χτυπήσουμε και την γραφειοκρατία και την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει πολλές από τις κινήσεις μας και κυρίως πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση των αναγκών. Ε, πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια αναπροσαρμογή της στρατηγικής ξεκινώντας από τη δημιουργία βασικών υποδομών στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης. Και έχουμε δει πολλά παραδείγματα όπου όταν ξεκινήσαμε από αυτούς τους δύο τομείς υπήρξε ραγδαία και δραματική ε, εξέλιξη και πρόοδος. Ε, για παράδειγμα, έχω ακούσει πολλές φορές να λέγεται για ένα αγωγό οπτικών ινών που θα καλύψει όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Ε, αυτό δεν είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει στην Αφρικανική Ήπειρο. Είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να κατασκευάσουμε πριν φτάσουμε στους αγωγούς οπτικών ινών που σε τελική ανάλυση δεν είναι και πάντοτε ό,τι καλύτερο για την δημοκρατία. Τέλος, όσον αφορά την, ε, τις κλιματολογικές αλλαγές, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η αναπροσαρμογή της στρατηγικής μας με βάση τα νέα δεδομένα και όχι να προσπαθήσουμε τώρα μέσα από την αναπτυξιακή βοήθεια να αλλάξουμε το κλίμα. Έχουμε κάποια δεδομένα, στη βάση αυτών των δεδομένων θα πρέπει να προσαρμοστεί και η βοήθεια. Κάποιες πρώτες παρατηρήσεις για αυτό το ζήτημα θα επανέλθω αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ για την ε, έκθεσή σας και για την ε, παρουσίαση και συμφωνώ ότι το Μπουσάν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, πολιτική μας συνολικά και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί ακουστεί με ενιαία φωνή, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπω προς το παρόν. Ίσως όμως τα πράγματα προχωρήσουν, ίσως το Συμβούλιο ε, δώσει κάποια όθηση, κάποια προσπάθεια καταβάλει. Επίσης υπάρχει και θέμα επίκρισης των δωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια. Ήδη τις προηγούμενες μέρες τα συζητήσαμε για την αποτελεσματικότητα. Και έχουμε όλες αυτές τις αρχές, όλες αυτές, όλες αυτές τις, τα συνθήματα για το, το value for money, να πιάνουν τόπο τα λεφτά, αυτό, γιατί αυτή την αυτοδιάδεση, την ιδιοποίηση, τη δημοκρατική, όλα αυτά, την ευθύνη, την υπευθυνότητα, όλα αυτά για την διακυβέρνηση σε αντισόμενες χώρες, όπου συμμερίζονται και αναλαμβάνουν κάποιο κομμάτι τη ευθύνη, αλλά ένα κομμάτι μόνο. Άρα συνεχίζονται οι επικρίσεις. Όσον αφορά το τι κάνει η Κομισιόν, τι κάνουν οι δικές μας κυβερνήσεις. Άρα θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στην αρχική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα όπως διατυπώθηκε στο Παρίσι. Να στα είπατε και από το Global Health. Γι' αυτό, γι αυτό το ownership, τι πάει να πει, τι ορισμός μπορεί να δηθεί. Ναι, συμφωνώ ότι χρειάζεται έλεγχο από την κοινωνία των πολιτών, χρειάζεται έλεγχο από κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι αφύπαρκτο που είναι και αυτονόητο ένα δυόμενε χώρε τώρα, κάτι το οποίο επίση ε, έχει σχέση με το Μπουσάν. Ε, και εκεί έχουμε κάποιου εταίρου, οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν. Αλλά δεν θα πρέπει οι χώρε εκείνες να είναι πρόφαση για να ματιώνονται αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί. Να το δούμε επομένω καλύτερα το θέμα. Και αυτό, το να είμαστε δηλαδή εμείς πιστοί στην αρχή της αποτελεσματικότητας ενίσχυση είναι και υπέρ των χώρων εκείνων. Άρα χρειάζεται προσπάθεια και πολιτική βούληση από όλου. μα. Συμφωνώ με τη μη κυβερνητική οργάνωση Action for Global Health για όσα μας είπατε. Ότι δηλαδή δεν τελειώνει η υπόθεση με αυτή την έκθεση. Πρέπει να χρειάζεται συνέχεια προσπάθεια, πίεση για να πετύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορτές. Σύντομο, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρέντα για την έκθεση και για το Action for Global Health θέλω να πω αυτό όσον αφορά αυτή το διαρθρωμένο χώρο για την κοινωνία των πολιτών. Όταν μιλάμε για τέτοια κοινότητα των πολιτών, εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι το οποίο είναι θολό, δεν είναι πολύ σαφές, ρευστό. Οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Συνδικάτα δηλαδή. Ενώσει φορείς ε, επιχειρηματιών, εργοδοτών. Όμως δεν είναι όλοι αυτοί οι φορείς αναγνωρισμένοι και ταυτισμένοι την έννοια της κοινωνίας των πολιτών, όπως ας πούμε λέμε για την ε, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Άρα, εάν υπάρχει τέτοια διάρθρωση, τέτοια δόμηση της κοινωνίας των πολιτών, αυτοί θα βγουν κερδισμένοι. Άρα θα πρέπει να ψάξουμε, να ξεκαθαρίσουμε περισσότερο αυτή την ιδέα για την κοινωνία των ε, πολιτών. Το, το λόγο τώρα θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως πάντα να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επικροτούμε την έκθεση. Σημαντική συμβολή αποτελεί για την προετοιμασία μας για τον Μπουσάν. Όσον αφορά αυτά που είπατε για τα αποδεικτικά στοιχεία, συμφωνούμε. Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι γίνονται αργές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε αποτελέσματα, προοδεύουμε πολύ αργά. Πώς πιστεύει η Κομισιόν ότι θα ενισχύσουμε την υλοποίηση στο μέλλον. Δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν, συμπληρωματικοί. Πρώτον, δεσμευόμαστε με τις δηλώσεις του Παρισιού και την ατζέντα της Άκρα για δράση πρέπει να προσδιορίσουμε προτεραιότητες και δράσεις που σχετίζονται με αναπτυξιακά αποτελέσματα. Πολλά ζητήματα έχουν αναφερθεί εδώ. Δημοκρατική αυτοδιάθεση, διαφάνεια και προβλεψιμότητα, καταμερισμός και καταλογισμός ευθυνών για τα αποτελέσματα. Προτεραιότητες για το μέλλον όλα αυτά για να ενισχύσουμε επίσης την ε, ατζέντα της ε, αποτελεσματικότητας ε, έχουμε δύο στοιχεία. Η υλοποίηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της αρρωγής είναι σημαντική για να επιτευχθούν αποτελέσματα και εξαρτάται από τη χρηματοδότηση διαφόρων ODA. Κατά την άποψή μας, Πρέπει να επεκτείνουμε τις αρχές αποτελεσματικότητας της αρρωγής σε διαφορετικούς τόπους χρηματοδότησης όπως καταπολέμησης της ε, κλιματικών αλλαγών, ιδιωτικές ε, επενδύσεις και τριγωνική συνεργασία. Οι αρχές λοιπόν αυτές ε, εδώ προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται επίσης να εμπλακούν περισσότερο οι διάφοροι εταίροι στην αποτελεσματικότητα της αρρωγής, ειδικότερα οι αναδυόμενες οικονομίες. Και η δική τους ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν πρέπει να μειώνει τις δικές μας φιλοδοξίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αρρωγής. Πιστεύω ότι η έκθεση σωστά επικεντρώνεται σε επίπεδο χωρών και προτείνει ευελιξία σε τοπικά πλαίσια. Υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι οι μελλοντικέ προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν σε επίπεδο κρατών. Κυρία Σρό, είχατε κάποια ερώτηση. Σας προτείνω λοιπόν να απαντήσετε στον κύριο Κόρτες. Κορτές. Έχετε ένα λεπτό. Ο ορισμός ενός ενθαρρυντικού περιβάλλοντος ε, συμφωνώ με την Κομισιόν για να συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών αυτό πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο θέλουμε να συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στο Σαλβαντόρ για παράδειγμα υπάρχει ένα φόρουμ όπου όλοι αυτοί μπορούν να συζητήσουν και να, δώσουν, ε, να συμμετέχουν σε ένα εθνικό σχέδιο. Ένα άλλο παράδειγμα για τη διάρθρωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ε, ένας μηχανισμός συντονισμού κρατικός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων, των χορηγών και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι εκλέγονται σε αυτές τις θέσεις και δίνουν πολύ χρήσιμα σχόλια για το πώς μπορεί να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέντα. Σας ξαναδίνω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Δύο λεπτά. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι σχολίασαν τα πράγματα τα οποία θα λάβω υπόψη και είμαι πεπισμένος ότι όταν συζητήσουμε τις τροπολογίες θα βελτιώσουμε την έκθεση. Επίσης, έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο λεπτά. Για πέστε μας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται όσον αφορά την ανακοίνωση που ε, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε την απάντηση, Κομισιόν, ναι. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο ίμιση του Σεπτεμβρίου θα εκδώσουμε την ανακοίνωση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κι άλλο χρόνο, αν θέλετε, ένα λεπτό. Σας το χαρίζω, κύριε Πρόεδρε. Τέλεια, τέλεια, λέει Πρόεδρος. Ωραία. Και Τώρα θα προχωρήσουμε στην ανταλλαγή των απόψεων με τον δόκτωρα Μπαμπατούντε όσο τι με είναι. Συγγνώμη που ε, προφέρω λάθος μάλλον το όνομά σας που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τον πληθυσμό. Και επίσης αναπληρωτής γραμματέας του ΟΗΕ. Μπορείτε να έρθετε να καθίσετε στο πλάι μου αν θέλετε και θα μας ε, μιλήσετε για αυτή την εντολή που έχετε για τις ε, πρόσφατες δράσεις σας και για τα σχέδιά σας. Alors, donc, et Madame Essenecker, la chef du bureau donc, de Bruxelles. του, του γραφείου της του της το Thank you very much, Madam Speaker. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σχετικά με την ε, Επιτροπή ε, Ανάπτυξης θέλω να σας χαιρετήσω όπως να χαιρετήσω και τους συναδέλφους και φίλους. Καταρχήν Χαίρομαι που με καλέσατε να σας μιλήσω διότι το προηγούμενο μήνα είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Αιθιοπία και στην Νιγηρία μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Μπάνκι Μουν και αυτό ήταν στα πλαίσια ενός ε, μιας περιοδίας για να ενισχύσουμε την ε, συλλογική στρατηγική εφόλης της ύλη και με αυτή τη στρατηγική αποβλέπουμε να σώσουμε τη ζωή 15 εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών μέχρι το 2015 που είναι ο στόχος για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, και ε, η εικόνα που είδαμε και η φωτογραφία που βλέπετε είναι στο επίκεντρο αυτού του οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε διότι εις ε, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τους λαούς ε, πρέπει να ε, δούμε ποιοι χρήζουν περίθαλψης, πού κατευθυνόμαστε και ε, πότε είναι έτοιμο, ε, θα είμαστε έτοιμοι. Διότι σαν ε, άνθρωποι πρέπει κανείς να μπορεί να έχει την ελευθερία επιλογής, σε ευκαιρίες. Οι γυναίκες πρέπει να δημιουργήσει την οικογένειά της όπως επιθυμεί, να μπορεί να γεννήσει ασφαλώς, χωρίς περιπλοκές να επιλέξει πότε θα κάνει παιδιά, τα παιδιά αυτά να ζήσουν ελεύθερα, χωρίς ε, AIDS και ε, να έχουν μια παραγωγική και επικοδομητική ζωή. Ε, διαβλέπουμε μια γενιά νέων οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, θα είναι πληροφορημένοι, θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα έχουν ευκαιρίες για να μπορέσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας επικοδομητικά. Εδώ μιλάμε για άνδρες και γυναίκες οι οποίοι πρέπει να αποδεχθούν τις ευθύνες ε, των ενηλίκων και να αφήσουν πίσω τους την παιδική ε, ε, στην κατάλληλη στιγμή, πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχουμε πετύχει σαν στόχο, διότι το 1994 είχα πάει στο Κάιρο για την ε, ιστορική διάσκεψη που είχε γίνει για την ανάπτυξη και τους πληθυσμούς και ε, όπου 179 λαοί είχαν συμφωνήσει να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δυνατότητα των ε, γυναικών να μπορέσουν να διαμορφώσουν τις επιλογές τους. Είχαν συμφωνήσει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα ε, ε, αναπαραγωγικής υγείας και καταλήξαμε σε μία κατάσταση, σε μία διαπίστωση ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη, αλλά το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Οπότε, όπως βλέπετε, στην επόμενη διαφάνεια παρόλες τις ε, προσπάθειες της ε, ε, διεθνούς κοινότητος 40% των χωρών ανά τον κόσμο ακόμη δεν έχουν επιτύχει τους στόχους να έχουν το επιτύχει στο MDG 5 για την υγεία της μητέρας και ο χρόνος πλέον εκπνέει διότι είμαστε ήδη στο 2000 2011 και ο στόχος μας είναι το 2015. Αρκετά χρόνια μετά από την κατάρτιση του MDG 5 που αναφέρεται στην ε, ε, παγκόσμια πρόσβαση σε αναπαραγωγική υγεία ε, καταρτήσαμε τον στόχο τον οποίο επιζητούμε ακόμη σήμερα διότι βλέπουμε ότι ακόμη πολλές γυναίκες πεθαίνουν κατά την διάκαιρη της εγκυμοσύνης ή της γέννας και υπάρχουν 15 εκατομμύρια γυναίκες που θέλουν να αποφύγουν τις εγκυμοσύνες χωρίς όμως να έχουν ε, πρόσβαση σε σύγχρονα αντισυλληπτικά μέσα. Και ε, εδώ δεν είναι μόνο αριθμοί και ε, στοιχεία, αλλά είναι προκλήσεις για να βοηθήσει κανείς τις γυναίκες. Το MDG 5 δεν έχει προχωρήσει όσο άλλα παρεμφερή προγράμματα και δεν υπάρχει μία συνεκτική και συλλογική δράση επί του θέματος. Θα θέλαμε ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για αυτό το MDG, πράγμα το οποίο αναγνωρίστηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο εις ε, την ε, ε, διάσκεψη που έγινε για τη δεκαετία της καταρτήσεως των προγραμμάτων αυτών, των MDGs και η αποτυχία ενός προγράμματος αποτελεί κίνδυνο και για τα υπόλοιπα. Χρειαζόμαστε στόχους και θα πρέπει οι στόχοι να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ενήλικες αλλά και τους νέους και εδώ βλέπετε ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για τους νέους διότι θα δείτε ότι ε, ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα διότι 90% των νέων ζουν σε υποανάπτυξη χώρες οι πληροφορίες σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι απαραίτητα και οι νέοι αυτοί ε, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της επομένης ε, γενιάς και αν δεν τους αντιμετωπίσουμε και δεν τους βοηθήσουμε τώρα δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και ε, το, ε, την αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίω πρέπει να έχουν δικαίωμα προσβάσεως εις ε, την, εκπαίδευση και την ενημέρωση και στην επόμενη διαφάνεια ε, ε, αναφέρουμε τι πρέπει να περιλάβουμε κατά τρόπον ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας εις, ε, τα, στους νέους αυτούς διότι όσο προχωράμε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι νέοι και η ανθρωπότητα κινδυνεύουν και έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή ε, να κινηθούμε διότι έχουμε ε, πάρα πολλά θέματα να επιλύσουμε την ε, επιστημιστική ασφάλεια, τις κλιματολογικές αλλαγές και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και ευκαιρίες πέραν των προκλήσεων. καθώς ο κόσμος θα φτάσει τα 7 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο, θεωρούμε ότι αυτός ο πληθυσμός θα αποτελέσει καταλήτη για να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα. Σήμερα είμαστε πιο αλληλοσυνδεδεμένοι από ποτέ, με περισσότερη ενημέρωση και περισσότερους πόρους και την ικανότητα να ξεπεράσουμε τα σύνορα και να βελτιώσουμε τις ζωές όλων στον κόσμο με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, με βελτίωση των ζώων όπου τα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν παιδιά. Για να ζήσουμε όμως μαζί σε έναν υγιή πλανήτη θα πρέπει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα σε ένα κόσμο 7 δισεκατομμύριων ανθρώπων θα πρέπει να υπολογίζουμε ο ένας τον άλλο υποστηρίζοντας τα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στις ε, αναπορικές τους επιλογές ε, δίνοντάς τους τις σωστές ευκαιρίες μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές επεκτείνοντας ε, της ε, πρόσβαση στη βοήθεια για την αναπαραγωγή θα καταπολεμήσουμε την παιδική θνησιμότητα και τη θνησιμότητα των μητέρων. Τα κοινωνικά ωφέλη και τα οικονομικά ωφέλη είναι προφανή. Ας μιλήσω λίγο για τους νέους. Από τα 7 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι και σχεδόν το 90% ζει στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εάν δεν αναλάβουμε δεσμεύσεις προς αυτούς με προενεργό τρόπο, ώστε να τους παρέχουμε ενημέρωση, εκπαίδευση, πρόσβαση σε αναπαραγωγική υγεία και υπηρεσίες αναπαραγωγικές, ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές. Αυτοί θα μπορέσουν να καθορίσουν την ανάπτυξη του πληθυσμού. Αν εξετάσουμε τα δημογραφικά στοιχεία παγκοσμία στον, στον αναπτυγμένο κόσμο, βλέπουμε ότι ο πληθυσμός είναι σταθερός ή μάλλον συρρυκνώνεται σε ορισμένες ανεπτυγμένε χώρες, ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο κλιμακώνεται αυξάνεται σε τερα... με τεράστιο ρυθμό και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάπως. Πρέπει να παρέχουμε πρόσβαση, εκπαίδευση, σεξουαλική εκπαίδευση, πρέπει να είμαστε να φροντίσουμε να τους παρέχουμε τα αγαθά τα οποία θα φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να κάνουν αυτοί έξυπνα τις σωστές επιλογές, ώστε ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος. Θα πρέπει να επενδύσουμε στον οικογενειακό σχεδιασμό και να μειώσουμε τη θνησιμότητα στις μητέρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. θα πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τις ε, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες να μειωθεί ο αριθμός τους, θα πρέπει να φροντίσουμε οι πόροι να ε, καταλήγουν στην φροντίδα για τις μητέρες και για τα παιδιά. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία ε, θα φέρει τα σωστά αποτελέσματα. Πάνω από τα δύο τρίτα έχουμε καταφέρει να τις συρρυκνώσουμε αυτές τις ανεπιθύμητες ε, και Έχουμε ένα πρόγραμμα συνεργασίας που ακόμα βέβαια πολλά θα πρέπει να γίνουν και η Γενική Συνέλευση παρέτεινε την, ε, το, το πρόγραμμα αυτό. Αύριο θα γίνει, του χρόνου θα γίνει αυτή η διάσκεψη του 20 συν και, έτσι θα διατυπωθούν κάποιες νέες προτάσεις. Ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αναπτυγμένος κόσμος θα βοηθήσει τις οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών, ούτως ώστε αυτός ο πληθυσμός των νέων θα βοηθήσει στην πρόοδο μέσα από την πράσινη οικονομία. Οπότε όλοι θα βγουν κερδισμένοι οικονομία, η ανάπτυξη, θα εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι θα γίνει ένας καλύτερος κόσμος, καλύτερος πλανήτης για τα παιδιά. Αυτό έχει σχέση με την αύξηση του πληθυσμού όπου έχουμε ως τώρα τους περισσότερους νέους από όσο ποτέ. Υπάρχουν επομένω εδώ τρεις κατευθύνσεις που θα κινηθούμε, εθνική ικανότητα ε, για τα συστήματα υγείας, δηλαδή θα πρέπει επίσης να τα βελτιώσουμε, υπηρεσίες για αναπαραγωγική υγεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ε, πρόνοια, την φροντίδα της υγείας, ε, επίσης ε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Χρειάζονται επίσης ε, προσωπικό, ιατρικό. και προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού. Πρόληψη και θεραπεία για το AIDS και αυτό να γίνεται σε κάθε επίπεδο παντού. Θα πρέπει να βοηθηθούν και οι εθνικές κυβερνήσεις ούτως ώστε μέσα στην ίδια του τη χώρα να βελτιώσουν τα πράγματα και έτσι οι πρωτοβουλίες για την ε, αναπαραγωγική υγεία να υλοποιούνται, να βοηθήσουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις με προγράμματα κατά τη ε, σεξουαλική βίας, του κοινωνικού προγραμματισμού και επίσης θα πρέπει να κινητοποιήσουμε οι ε, οικονομικούς πόρους. Γιατί σήμερα με τα τελευταία στοιχεία έχει υπάρξει σταθεροποίηση γύρω στα 10 δις δολάρια ετησίω όσον αφορά αυτά τα προγράμματα. Ε, λόγω της κρίσης βέβαια δεν πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις. ένα δις ετησίω για τις σχετικέ δραστηριότητε. επίσης έχουν κινητοποιήσει οι χώρες χώρε, αλλά χρειάζονται περισσότερα ε, βοήθεια από τους δωρητές. Αν, αν συνεχιστεί θα έχουμε 24 δις λιγότερα από ό,τι χρειάζεται για να χρηματοδοτήσουμε τα πρόγραμματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πρωτοπόρα η Ευρώπη, είναι γνωρισμένη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το έναν δις που θα πρέπει ο κ. Μπαρόσο να φροντίσει να δοθεί, ιδίως για ε, την υγεία των μητέρων. Πάρα πολύ σωστή αυτή η πρωτοβουλία και ως Ένωση, ως Κομισιόν θα πρέπει να πούμε σε όμως χώρες ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν αρκεί, θα πρέπει να κοιτοποιήσουν και τους δικούς τους πόρους. βοηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά αυτό το οποίο θα στηρίξει την πολιτική αυτή είναι η εθνική πόρη. Και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει σε διμερείς εννοήσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις. Έχουμε αντιλησχίσει με συμπεράσματα όσον αφορά καινοτόμε λύσεις που όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Να επενδύσουμε στην ε, ε, αναπαραγωγική υγεία, χρονικό προγραμματισμό και θα πρέπει αυτά να γίνουν υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές μας. Η Ευρώπη να συνεχίσει και να αναβαθμίσει την εξωτερική δράση προς αυτή την κατεύθυνση. δικαιώματα των γυναικών, εκρίζωση τη φτώχειας και βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Αυτό χρειάζεται να γίνει σε όλους σε αυτούς που είναι στο περιθώριο και θα πρέπει στη συνεργασία με τους ε, εταίρους μας αυτά όλα τα θέματα να τα εντάξουν σε όλες τις πολιτικές, θέματα για τον πληθυσμό, για τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα πολιτικής που έχουμε και τώρα. Για να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Θέλω να σας δείξω ότι στο UNFPA εστιαζόμαστε στην καρδιά της ατζέντα του ICPD. Στο UNFPA θέλουμε να προάγουμε την ε, αναπαραγωγική υγεία, να μειώσουμε τη θνησιμότητα των μητέρων, και να επιταχύνουμε την πρόοδο στην ατζέντα του ICPD και για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, ώστε να βελτιώσουμε τις ζωές των πληθυσμών, ειδικότερα των γυναικών, των νέων και των εφήβων. Δίνοντας τους, ε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τη δυναμική του πληθυσμού και η UNFPA είναι ο μόνος οργανισμός που έχει πρόσβαση και διαχειρίζεται δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης μας απασχολούν. Ο UNFPA βρίσκεται σε 29 χώρες και συνεργάζεται με εθνικά συστήματα. Συνεργαζόμαστε με εκατοντάδες οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεις από ολόκληρο τον κόσμο, οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, και ε, είμαστε, χρησιμοποιούμε το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ε, βασίζεται στη συνεργασία. Χαιρόμαστε για τη συνεργασία μας με τους μη οργανισμούς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα Ηνωμένα Έθνη επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να φέρουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο επίπεδο για τους κοινούς στόχους προς το κοινό καλό για μεγαλύτερο και πιο βαθύ πολιτικό διάλογο. Τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτευξή αυτών των στόχων. Πριν ε, ολοκληρώσω θα σας δείξω αυτό, γιατί αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύω ότι το όραμα του UNFPA για υγιείς και ενδυναμωμένες γυναίκες, έφηβες ε, κοπέλες και νέους ανθρώπους είναι κάτι που δύσκολο, αλλά συνεργαζόμενοι μαζί σας και δεσμεύοντας τους απαραίτητους πόρους μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το όραμα. Εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο για την εκπλήρωση αυτού του οράματος. Έχουμε την ικανότητα να επρασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών, των έφηβων κοριτσιών και των νέων ανθρώπων μέσω δράσεων και αποφάσεων να, αποφύγουμε, να βοηθήσουμε τις ζωές των γυναικών και των εφήβων σε ολόκληρο τον κόσμο και να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών ώστε οι πληθυσμοί να είναι υγιείς και οι εγκυμοσύνες να είναι όλες επιθυμητές. Πληθυσμός δεν σημαίνει μόνο νούμερα. Πληθυσμός σημαίνει ανθρώπους. Σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημιουργία συνθήκων, ώστε όλοι να ζουν σε έναν υγιή πλανήτη και να ε, μπορούν ε, να ε, εφαρμόσουν, τις, να υλοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Μπορούν, πρέπει να μετράμε, να υπολογίζουμε όλοι ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική, ε, για την εξαιρετική παρουσίαση και το λόγο έχουν τώρα οι βουλευτές. Ξεκινάει ο κύριος Κάσμαν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, δόκτωρα, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Έχασα τα δύο πρώτα λεφτά μεν διότι απουσίαζα, αλλά ήταν εξαιρετική και συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε. Είμαι ο εισηγητής του Κοινοβουλίου σχετικά με την επίτευξη των ε, στόχων της χιλιατηρίδας και είχα συμμετάσχει στην διάσκεψη όπου ο πρόεδρος Μπαρόζο δέσμευσε ακόμη ένα δισεκατομμύριο για τους στόχους αυτούς. Όντως η θνησιμότης των γυναικών και των παιδιών είναι ε, βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών. Οπότε συμφωνώ μαζί σας. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω ήταν ε, να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου διότι όλοι σε αυτό το κοινοβούλιο δεν συμφωνούν με τις προσεγγίσεις ε, που διατυπώσατε εσείς ή αυτά που λέμε εμείς. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας, διότι ορισμένοι θεωρούν ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είναι ο εχθρός της γυναίκας, ενώ είναι ο εχθρός της καταστολής και της καταπίεσης και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι είναι βασική η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σεβαστούμε τις επιλογές και τονίζω τη λέξη επιλογές δουλειές τις οποίες ε, κάνουν οι γυναίκες διότι όλες οι ε, ε, αποτυχίες μπορούν να αποφευχθούν. Πρέπει λοιπόν να καταργήσει κανείς την πολιτική, να επικεντρωθούμε στις ανάγκες του διότι ε, υπάρχουν γυναίκες και παιδιά που κινδυνεύουν λόγω της γένας. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια συλλογική ε, προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ δεν κοιτούν ίσως τα προβλήματα επιτόπου όπως στην Ποτσουάνα όταν πηγαίνω όπου εν τρίτον του ΑΕΠ ε, διατίθεται για την ε, πρόληψη και την καταπολέμηση του AIDS. Ε, όταν λοιπόν κοιτάζουμε τα προβλήματα αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην πραγματικότητα και βλέπουμε την εργασία που γίνεται στην την Νότιο Αφρική. Βλέπουμε πόσες γυναίκες που έχουν θετικό ιό του AIDS αλλά δεν μεταφέρουν πια τον ιό αυτό στο παιδί τους λόγω ε, παιδείας, λόγω πληροφόρησης. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και που πρέπει να κάνετε και εσείς για λογαριασμό μας είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσετε ότι θα συμβάλλουν τον στόχο τους για την αναπτυξιακή βοήθεια βοήθεια και ε, να ε, εξασφαλίσουμε και τις επιπρόσθετες ε, χρηματοδοτήσεις που είναι αναγκαίες για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν ήταν υποχρέωση, ήταν μία προσπάθεια, μία φιλοδοξία και τώρα εφόσον έχουμε δεσμευτεί πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας. Ευχαριστώ για το θαυμάσιο κείμενό σας. Ε, είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα. Ε, εξηγεί την δουλειά σας ε, και των άλλων οργανισμών και θα το χρησιμοποιήσω αλλά χωρίς τη βοήθεια των άλλων δεν θα μπορέσουμε να επιτρίχουμε τίποτα διότι υπάρχει μία μάχη την οποία μάχη πρέπει να είμαστε πολλοί για να την κερδίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Το λόγο λόγο έχει η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να σας πω ότι μερίζομαι, ότι συμμερίζομαι το όραμά σας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχω δουλέψει με οργανισμούς που συνεργάζονται μαζί σας και έχω ιδίαν εμπειρία για το τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω από κάτι που το έχω ξαναπεί. Η βιολογία έχει τους δικούς της κανόνες και αυτή η αύξηση του πληθυσμού της γης υπακούει σε κάποιους κανόνες και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν ρυθμίσουμε εμείς την αύξηση του πληθυσμού, η ίδια η φύση θα το ελέγξει όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και καμιά φορά το ρυθμίζει με έναν τρόπο που δεν μας αρέσει καθόλου. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί οργανισμοί σε επίπεδο μη κυβερνητικών που δουλεύουν και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απολαμβάνουν τη στήριξη της κοινωνίας όπως άλλοι οργανισμοί γιατί ακριβώς ο στόχος τους δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Συνεπώς, όπως έχω πει και άλλες φορές, πρέπει να γίνει η επανεκπαίδευση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τόσο ώστε να κατανοήσει και ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός τι σημαίνει ακριβώς σεξουαλική αγωγή, αναπαραγωγικά δικαιώματα, ε, αγωγή υγείας και όλα τα συναφή. Και επιπλέον χρειάζεται μια αυξημένη οικονομική στήριξη προς αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν την στήριξη της, ε, της κοινωνίας. Το επόμενο που θέλω να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλά λάθη. Για παράδειγμα, η ε, αναπαραγωγική υγεία έχουμε δει πολλές φορές να περιορίζεται στη διανομή των προφυλακτικών σε τεράστιους πληθυσμούς και βλέπαμε την άλλη μέρα τα προφυλακτικά στα χέρια των παιδιών να τα φυσάνε σαν παλόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικό. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που έχετε πει σε κάποια αποστροφή της ομιλίας σας. Από την αγωγή υγείας, από την σεξουαλική αγωγή, από την εκπαίδευση στα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Γιατί χωρίς αυτά μέσα σε ένα ε, παγκόσμιο πόλεμο εναντίον της φτώχειας δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ε, τις λύσεις για τα επιμέρους ε, προβλήματα. Ναι, είναι απαραίτητα τα σύγχρονα αντισυλληπτικά μέσα. Είναι απαραίτητο να σταματήσουμε τη μετάδοση του ιού από τις μητέρες στα παιδιά και βεβαίως να με συγχωρέσει ο φίλος μου Μάικλ uh, Κάσμαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με την εκπαίδευση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει χορήγηση φαρμάκων, τα οποία για την ώρα κοστίζουν πολλά λεφτά αλλά με τις ινδικές προδιαγραφές, όπως έχει ανακοινωθεί πρόσφατα, με 2 έως 9 δολάρια μπορεί αυτό να επιτευχθεί και δεν είναι τρομακτικό ποσό τα 2 με 9 δολάρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των εκτρώσεων. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει, που να μπορεί να απαγορεύσει ή νόμος που να καθιστά νόμιμες ή μη νόμιμες τις εκτρώσεις. Η κάθε μία γυναίκα μπορεί να αποφασίσει μόνο για τον εαυτό της. Και από τη στιγμή που θα αποφασίσει να προχωρήσει σε έκτρωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ασφαλή έκτρωση. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε για όλο τον κόσμο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του mutilation. Βεβαίως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά πολλές φορές το ξεχνάμε γιατί έχει περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Αφρικής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ε, βιασμούς και πάνω απ' όλα πρέπει να διδάξουμε τον κόσμο πώς να απολαμβάνει τον εαυτό του χωρίς να κινδυνεύει από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κέλλερ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Λέτε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι έτοιμες να παντρευτούν όταν είναι έτοιμες σώματι και ψυχή. Και επίσης ε, θα προσθέσω ότι πρέπει να είναι ελεύθερες να παντρευτούν όποιον θέλουν, ακόμη και αν θέλουν να παντρευτούν μια γυναίκα. Και να μην δίνουν λογαριασμό σε κανένα, διότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο σύζυγοι, δεν είναι μόνο μητέρες, παρότι συχνά οι μητέρες είναι γυναίκες, ε, οι γυναίκες δεν είναι πάντα μητέρες και πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτω φυσιολογικό. Θα ήθελα επίση να συζητήσω για τον αναπτυξιακό στόχο τη χιλιετία 5. Μου φαίνεται αστείο ότι αποτυγχάνουμε περισσότερο σε αυτό το στόχο. Η μείωση της φτώχειας φυσικά είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα, παραγωγή, παρα... ποιος παράγει τι, αλλά η υγεία για τις μητέρες αφορά περισσότερο την παροχή υπηρεσιών υγεία, εκπαίδευση. Ξέρουμε όλοι πως γίνεται, δεν υπάρχουν μεγάλε διενέξει όπω ε, για την καταπολέμηση τη στόχια. ωστόσο δεν επιτυγχάνουμε του στόχου. Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως ε, δεν λαμβάνει την απαραίτητη πολιτική προσοχή, φαντάζομαι. Ποιο είναι το πρόβλημα ουσιαστικά, είναι θέμα χρηματοδότησης, ε, είναι θέμα... Ποιο είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά το οικογενειακό προγραμματισμό, συμφωνώ με τον κύριο Κάσμαν. Όπως φέρεται η πλειοψηφία, συμφωνούμε σε αυτό. Ο προγραμματισμός είναι μια χαρά, αλλά πολύ συχνά ορισμένα πράγματα δεν προγραμματίζονται, όπως η βία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν προγραμματίζονται και ο προγραμματισμός μερικές φορές μπορεί να αποτύχει. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε στις περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει ή είναι αδύνατος ο προγραμματισμός διότι οι γυναίκες δεν είναι πάντοτε ελεύθερες να επιλέξουν τις σεξουαλικές τους δραστηριότητες και συμφωνώ ότι κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να είναι επιθυμητή και απέχουμε δυστυχώς πολύ από αυτό. Και αυτό λοιπόν το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ο προγραμματισμός είναι σημαντικός αλλά δεν είναι πανάκια. Η ερώτησή μου όμως είναι συγκεκριμένη διάφοροι άνθρωποι πιέζουν την Κομισιόν, αλλά για ποιο, ποιο, ποιο είναι το πρόβλημα. Το λόγο έχει ο κύριος Κόρτες. Sí, señor Rosetimen. en primer lugar lo que quería es felicitarle porque, <clears throat> por su intervención y sobre todo porque comparte. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα είπατε και όπως είπε ο κύριος Κάσμας. η πολιτική μας ομάδα συμφωνεί ως επιτοπλίστων με τον ε, ομιλητή μας. Πέστε μας τη γνώμη σας. Σας άκουσα, θέσατε κάποια προβλήματα. Εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα αυτά τα οποία, ε, προς, αυτά στα οποία προσκρούει το έργο σας για να μην μπορεί να πετύχετε τους στόχους σας. Εδώ συζητούμε πάρα πολλά. Όχι μόνο για τις σχέσεις με κυβερνήσεις, μιλούμε και για προβλήματα ιδεολογικά, προβλήματα θρησκευτικά, για πάρα πολλά ζητήματα ουσίας. Τα οποία φαντάζομαι και εσάς εμποδίζουν από το να επιτέλεσετε το έργο σας. Οπότε, για πέστε μας, τι γίνεται με τους νέους που εσείς έχετε αναδείξει στις προτεραιότητά σας. Δεν θέλω να μιλάω για τη χώρα μου, αλλά ένα παράδειγμα είχαμε με ένα μια συνάντηση ε, το, τον Αύγουστο ε, που αφορούσε κάποιους νέους καθολικούς και έλεγαν εφημερίδες ότι ε, υπήρχε κάποια καταστολή της εκστρατείας που αφορούσε τη χρήση προφυλακτικών ε, Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα παντού, υπάρχουν ζητήματα γύρω μας τα οποία ζητούν λύσεις. Και επομένως αυτό πρέπει να δούμε τα πραγματικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Άλλο πρόβλημα που μας αναφέρατε. Έχουμε ένα ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτές τις αντιληψόμενες χώρες. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι όλοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι χρειάζονται υγεία, χρειάζονται παιδεία, ακριβώς όπως ανέφερε ο συνάδελφος και η συνάδελφη πριν. Και Πώς θα αντιδράσουμε τώρα, ε, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους νέους, κόβοντας πόρους για αυτές τις αντισόμενες χώρες. Αντί γι' αυτό, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ποντάρουμε σε αυτές τις χώρες. Εκεί έχουμε πάρα πολλέ αιστείε φτώχεια. Χρειάζονται εκεί πέρα παιδιά, χρειάζεται υγεία και να βοηθήσουν τόσο ώστε αυτέ οι χώρε να μπουν στο κλαμπ των αναπτυγμένων χωρών, στην κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών και να έχουμε βεβαίως ισόρροπη, ισορροπημένη παροχή στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πάρα πολλά μας είπατε, εγώ απλώς μερικά από αυτά που είπατε σχολίασα. Πρόεδρος Νέζερ και κατόπιν ο προσκεκλημένος μας θα ξαναλάβει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον προσκεκλημένο μας, αλλά επίσης έχω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε το εξή, Μιλήσαμε για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης προηγουμένως και το θέμα είναι ακριβώ πώ θα γίνει πιο αποτελεσματική η Γενική Διεύθυνση πέντε που ασχολεί με την υγεία. Και έχουμε κάποια παραδείγματα χωρών που μα δείχνουν ότι εκεί πιάνει το η βοήθεια. Άλλε χώρε αντίθετα δεν πιάνουν το 0,7%. Θα πρέπει νομίζω να αποκαλύψουμε ποιε είναι οι χώρες οι οποίε. Ε, τηρούν το στόχο του 0,7 και ποιες όχι. Να κατονομαστούν. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά τα στοιχεία, νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει. Α, ένα παράδειγμα είναι η Ουγγάντα. Ο πληθυσμός έχει φτάσει 30 εκατομμύρια. Τα έχει ξεπεράσει. σύντομα θα έχει πιο πολύ πληθυσμό αυτή η χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την εξαγγελθήσα πολιτική και το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα, όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το αξιότιμο ακροατήριο για όλα τα σχόλια που μου δίνετε. Τα σημειώνω και τα λαμβάνω πολύ σοβαρά. Θέλω να υπογραμμίσω ότι Ε, έχουμε θέσει ως στόχο, ως γρήγορο στόχο και μπορούμε να τον επιτύχουμε γρήγορα τη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί. Θα μιλήσω για κάποιους συγκεκριμένους που πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για ποιο λόγο δεν επιτυγχάνουμε τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας νούμερο 5, διότι το ζήτημα της νησιμότητας των μητέρων, των μητέρων είναι ένα πρόβλημα στο οποίο συμβαλούν πολλοί παράγοντες. Ορισμένοι εξωτερικοί από τον κλινικό χώρο, από το χώρο των ιατρών. Είναι πολιτιστικοί οι παράγοντες αυτοί. Σχετίζονται με τη θρησκεία, με την ε, καθεστώς των γυναικών και πρέπει να φροντίσουμε να συνεργαζόμαστε με τοπικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτούς, να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς με κατά κάποιο λόγο φύλακες οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις γυναίκες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ήμουν υπουργό Υγείας στην Ιγυρία. Είχαμε προβλήματα με τον εμβολιασμό και την πολιομιελίτιδα σε μια περιοχή της χώρας. Δεν είχαμε πρόσβαση στα παιδιά τα οποία έπρεπε να εμβολιαστούν. Και αυτό που χρειάστηκε να κάνουμε ήταν να συνεργαστούμε με θρησκευτικέ οργανώσεις σε εκείνο το μέρος της Νιγηρίας, ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την κοινότητα. Εντός ενός έτους μειώσαμε τον επιπολασμό κατά 90% για την πολιομελίτιδα επειδή συνεργαστήκαμε με τοπικές κοινότητες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη, να διαγιγνώσκουμε την ίδια την κοινότητα, να έχουμε ενδιαφερόμενους επί τόπου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ότι όπως είπα νωρίτερα, πρέπει να συνεργαζόμαστε με κρατικές υπηρεσίες τόπου ώστε να λαμβάνουν τις δύσκολες επενδυτικές αποφάσεις. Δεν έχει νόημα να επενδύουμε ε, στην άμυνα σε μια αναπτυσσόμενη χώρα όταν οι άνθρωποι πεινούν. αυτού είναι, αυτά είναι τα επιχειρήματα αυτού του είδους πρέπει να προωθήσουμε, πρέπει να οικοδομήσουμε τα συστήματα υγείας. Τελικά το σύστημα υγείας είναι σημαντικό ε, και δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία, είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων, είναι για να προσφέρει φάρμακα αλλά και για να προσφέρει υγεία προσωπικό φροντίδας είναι, ε, προορίζεται ώστε ο, ο υπεύθυνο για τη φροντίδα της κοινότητας να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει. Σε αυτές τις περιοχές θα διαδοθεί ιδιαίτερα ο οικογενειακός προγραμματισμός. Εάν γίνουν οι σωστές επενδύσεις, συνεργαστούμε με τις ε, τοπικές κυβερνήσεις και ίσως συγχρηματοδοτώντας αυτά τα αυτού στους στόχους μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν επιτευχθούν τα τελικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε τα προγράμματα. Το ζήτημα του αναπτυξιακού στόχου 5 αφορά ακριβώς αυτό. Τέλος, ε, ήθελα να τονίσω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε έτσι να ενοποιήσουμε σε επίπεδο πρωτεύουσας ε, πρωτεύουσων υπηρεσιών, πρωτεύουσων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες που παρέχουν ελέγχους και ενημέρωση για το HIV, ε, ελέγχους εγκυμοσύνης, ε, εμβολιασμούς, ε, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού. Αν τα κάνουμε και τα τέσσερα αυτά μαζί, μειώνουμε τη θνησιμότητα για τις μητέρες και για τα παιδιά. Άκουσα μια ερώτηση για τα, τα ζητήματα, ποια είναι τα προβλήματα που, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι προκλήσεις ε, σχετίζονται με την εντολή μας. Η εντολή μας, ε, η αποστολή μας ε, μιλάει για ζητήματα πολύ προσωπικά για τους ανθρώπους, για τις ανθρώπινες ζωές, για τους ανθρώπους. Υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχουν θρησκείες, υπάρχει ο πολιτισμός. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Πιστεύουμε ότι σε κάθε περιβάλλον θα πρέπει να μπορέσουμε να το αποδομήσουμε κατά κάποιο τρόπο και να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να το κατανοήσουμε. Επίσης, ε, όταν, όταν μιλάτε για την ικανότητα, για τη δυνατότητα των γυναικών να παντρευτούν όποιον και όποιαν θέλουν. Συμφωνώ με αυτό, αλλά στο πλαίσιο του αναπτυσσόμενου κόσμου, εάν δούμε πραγματικά τι συμβαίνει εκεί, τα νέα κορίτσια παντρεύονται στην ηλικία 12-13, δεν γνωρίζουν καν τι είναι. Τα σώματά τους δεν έχουν ακόμα οριμάσει, τόσο ώστε να γεννήσουν παιδιά δεν έχουν σε αυτή την ηλικία ούτε καν την αίσθηση του ποιε είναι. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λοιπόν της ηλικία γάμου, της πρόσβασης σε εκπαίδευση, της πρόσβασης σε υπηρεσίες. Αυτό είναι το ουσιώδες πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να μιλάμε. Ήθελα να πω ότι από πολλές απόψεις ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι Αυτές οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο. Ο, δεν βρίσκονται αυτές οι προκλήσεις εδώ στις Βρυξέλλες, ούτε στην Ευρώπη. Βρίσκονται σε τόπους όπου, όπως γνωρίζετε, στην Ποτσουάνα, στο Νεπάλ, στο Αφγανιστάν. Αυτά είναι τα μέρη στα οποία πρέπει να πάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλουμε τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν προγράμματα. Κάθε κράτος μέλος να έχει ένα εθνικό πρόγραμμα αντιμετωπίσεως αυτών των θεμάτων. Και εμείς σαν ΟΗΕ θα συγκεντρώσουμε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους για να κοστολογήσουμε τα προγράμματα και να ε, καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα εφαρμογής, να τους ε, δείξουμε τι μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη το Global Fund, το Παγκόσμιο Ταμείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να παρέμβει σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να χειροκροτήσουμε τον μιλητή και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών που είναι ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πρέπει να εξετάζουμε ε, τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών στις υποανάπτυξη χώρες και αναφέρομαι εδώ στις ε, κατά μέρους πολιτικές γεωργίες, βιομηχανίες, ανάπτυξη λοιπά. Η κυρία Σίμπερ Στάστραμ είναι η μόνιμη εκπρόσωπος της Επιτροπής μας η οποία θα μας παρουσιάσει ε, τα βασικά θέματα της εντολής της και ορισμένα βασικά, ορισμένες βασικές παρατηρήσεις για την ανάπτυξη, για την πολιτική μετανάστευση και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την παρουσία της και τον εκπρόσωπο που θα συμμετέχει. Κυρία Έστραμ, δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να είστε σύντομοι διότι οι διερμηνείς θα μας εγκαταλείψουν όσον ούπο. Κυρία Στίμπελ Ζάστρα, με έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, όντως θα είμαι ταχύτατη και θέλω να αφήσω τη δυνατότητα στη Λόρα Σάλιβαν να μιλήσει γιατί είναι το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει ήδη ένας αέρας θερινών διακοπών και στο Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της συνοχής των πολιτικών έχουμε καταρτήσει ένα δίκτυο με την Επιτροπή με μη κοινοβουλευτικέ οργανώσεις, με ευρωβουλευτές και βουλευτές εθνικούς κατά τρόπον ώστε να παρακολουθούμε κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, διότι οι δικές μας δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες. Ε, έχουμε μέχρι στιγμής άτυπες ανταλλαγές με άλλες επιτροπές και θα πρέπει να υπάρξει μία πιο επίσημη μορφή κατά τρόπον ώστε να υπάρχει συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και ε, σε άλλα θέματα στη χορήγηση πιστώσεων από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και υπάρχουν και μία σειρά εκδηλώσεων ε, και ε, γι' αυτό χαιρετίζω την κυρία Σάλιβαν που θα μας τις παρουσιάσει. Δεν θέλω εδώ να αναφερθώ ε, ή στις πρώτες ύλες γιατί η Επιτροπή υλε γιατι έχει διατυπώσει μία σειρά προτάσεων και γι' αυτό ε, θέματα τα οποία θα μπορούσαμε ίσως αυτονόητα εμείς να χειριστούμε χειρίζονται, ε, εξετάζονται σε άλλες επιτροπές και υπάρχει ήδη μία επαφή με την Τράπεζα Επενδύσεων και οι πιστώσεις ε, ελέγχονται και ε, θα υπάρξει μία επιστροφή. Ε, επιπλέον υπήρχαν δι άφορες άλλες προβληματικές διαθέσεις πιστώσεων στη Μαδαγασκάρη ε, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε αλλά δυστυχώς η Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταρτήσει μία μελέτη που είχαμε προτείνει σε αυτό το τομέα και αν ε, έχω ενημερωθεί σωστά ο κύριος Μπέρμεν το έχει ξανασκεφτεί και θα διατυπωθεί μία πρωτοβουλία διότι πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό. Είναι ένα σημαντικός χώρος ο οποίος χρήζει μεγαλύτερη σημασία ιδίω όσον αφορά την ε, μετακίνηση, ε, μετανάστευση και την ε, πολιτική συνοχή για να ελέγξουμε τις ροές των προσφύγων διότι για να έχει νόημα κάτι τέτοιο πρέπει να αναρωτηθούμε επί ενός άλλου βασικού θέματος που δεν υπολογίζεται επαρκώς την ε, μετακίνηση από νότο εις νότον που έχουμε υποτιμήσει μέχρι στιγμής. Υπήρξαν ορισμένες ε, ε, ε, ορισμένες κινήσεις. Ο κύριος Γκιόρενς, η κυρία Κέλλερ σήμερα θα οργανώσει μία εκδήλωση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αξίζει να την επισκεφθείτε. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε ε, για την, ε, ε, ε, για την αλλαγή κατευθύνσεως που μας απασχολεί επίσης το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών είναι τόσο τεράστιο ότι θα χρειαζόταν μια ιδιαίτερη συνεδρίαση μου ελέγχθη ότι δεν πρέπει να μιλήσω επιμακρών και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους που μας έχουν βοηθήσει και την κυρία Σάλιβαν η οποία θα λάβει το λόγο τώρα. Η κυρία Σάλιβαν, επομένω, έχει το λόγο. Πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Λόρα Σάλιβαν της Action Aid. Είναι μια οργάνωση ε, της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας. 50 αντιπροσωπείες ε, έχουμε διεθνώς για να κατανοήσουμε την φτώχεια. Σήμερα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο όπου δεν έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το οποίο δεσμεύτηκε να κάνει με τη Λισαβόνα. Ε, οπότε θυμάμαι ότι λέγανε ε, τι, τι, ακριβώς εδώ πέρα, τι, τι έχει σημασία, τα, τα βιοκαύσιμα, τα PCT, όχι και, και, και τα μεν και τα δε, είναι κάτι τεχνικό, είναι κάτι συγκεκριμένο ταυτόχρονα. Και θυμάμαι ότι μιλούσαμε για κάτι συσκευές επικοινωνίας, δεν τα βρήκαμε και τελικά αυτό το BCD δεν εμπνέει κανέναν. Τελικά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι θέμα δίκαιων πολιτικών. Επομένως αυτό που τώρα θέλω να κάνω είναι να σας μιλήσω γρήγορα για αυτή την περίπτωση ε, για ε, την ε, ασφάλεια ενεργείας σε σχέση με την σχετική οδηγία. Το 2008 είχαμε τον στόχο 10% για, να, για χρήση ανανεώσιμων πηγών με το 2020. Πάρα πολύ επενετό σαν στόχος, όμως ε, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη προτίθενται να καλύψουν αυτό το στόχο ε, μέχρι το 92% για αυτή την πρώτη γενιά των βιοκαυσίμων που απαιτούν πάρα πολύ γη για να παραχθούν στην Ευρώπη. Ε, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε τέτοιο, τόσο, τόσο, τόσο, τόσο γη και έτσι δεν μπορούμε να το κάνουμε για τα βιοκαύσιμα. Επομένως έτσι ετέθη το θέμα και είχαμε και κάποιες ε, εταιρείε που ε, έλαβαν υπόψη αυτούς τους ε, στόχους και επομένως προχωρούμε σε κάποιες περιοχές του κόσμου όπως την Κένια. Να, εδώ πέρα έχουμε αυτή την ε, περιοχή, Ντακάτσα λέγεται, ή στην ε, Κένια όπου γίνεται μια τέτοια προσπάθεια το 2008. Έχουμε μια εταιρεία Ιταλική, Νι Γιώτα και στην Τακάτσα 5.000 εκτάρια έχουν μισθώσει 5.000 ροντεμάχυλα. Ε, και οπότε ε, αυτό το, το πήραν κόψε χρονιά κάτω από την αγοραία τιμή. Ε, δεν δόθηκε καμιά αποσυζημίωση και θες απασχόλησης ε, ε, είναι άγνωστο η κάθε, το κάθε άλλο άλλων την εταιρεία και άρχισε αυτή η φοιτεία χωρίς να έχει δώσει το πράσινο φως από την κοινότητα και ήρθαν σε εμά ή της κοινότητας, ζήτησαν βοήθεια και εμεί προσφύγαμε στην κυβέρνηση για τον Ιούλιο του 2010 αποφασίσανε να αναβάλουν την προσπάθεια. Ζητήθηκε από την εταιρεία να επανυποβάλει αίτηση πιλωτικού προγράμματος για 10.000 εκτάρια. 20.000 είναι αυτοί οι οποίοι ζούσαν εκεί και εκεί ε, ε, ξυλία, τρόφιμα, όλα αυτά ε, τα πουλάνε και ζουν. Χρήσαν και ένα σχολείο με χρήματα της Ένωσης και θα πρέπει να γκρεμιστεί. Να λοιπόν γιατί αυτή η περίπτωση, η παρουσίαση μας είναι ενδιαφέρον. Επίσης βλέπουμε ότι σε δύο επίπεδα ασχολούμαι με αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και θέμα ευθύνης της κυβέρνησης της χώρας. Για να δούμε πώς δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Το δικαίωμα στη γη, το δικαίωμα ε, στα προϊόντα τους, όλα αυτά έχουν παραβιαστεί. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια από την κίνητρο και κάποιες εταιρείες να πάνε εκεί που υπάρχει φτηνή γη. Επομένως, ε, ε, ε υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, δεν φταίνε μόνο τα δύο καύσιμα. Ε, η Παγκοσμία Τράπεζα. Θεωρεί πάντως ότι από τέτοιου είδους εξαγορές γεών ε, ένα 20 με 30% οφείλεται στα βιοκαύσιμα. Μεγάλη πίεση υπάρχει όσον αφορά το ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, να παγώσουμε αυτούς τους στόχους μέχρι ότου μελετηθεί καλά ο αντίκτυπος. Όμως και εν εγκατακλείται σε σχέση με αυτό που συζητούμε σήμερα δεν αρκούν αυτά τα οποία έχουν γίνει γιατί χρειάζονται πλαίσια συγκεκριμένα συνοχή αντιξιακών πολιτικών και σε συνδυασμό με την πολιτική μετανάστευση, σε εμπορική πολιτική και έχουμε τρία πράγματα που ζητούμε και θέλουμε την προσπάθειά σας μέσα στους μήνες και χρόνια μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση για φυσική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει την υποχρέωση της Ένωσης Λισαβόνας για συνοχή ενωτησιακών πολιτικών. Αυτό είναι το ένα. Να υπάρχει πολιτική ηγεσία, ανάληψη ευθύνη στο υψηλό, ύψιστο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Μπαρόσο, δηλαδή και η κυρία Άστον και συντονισμό από τον κύριο Πίμπαλεξ, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο κύριος Πίμπαλεξ. Ε, χρειάζεται να το στήριξουν και άλλοι επίτροποι. Τελειώνω, τελειώνω. Επίσης, χρειάζεται η ικανότητα εφαρμογή της πολιτικής. Να στηρίξει το κοινοβούλιο, πιο πολύ ε, προσωπικό να υπάρχει και όχι μόνο για την ε, πολιτική ανάπτυξη. Επίσης χρειάζονται κάποιοι μηχανισμοί που να βοηθούν. Ξέρω ότι τα συζητάτε με την Concord τώρα. Συνεργαζόμαστε. Θα υπάρξει μια μελέτη τον Οκτώβριο. Θα καλύψουμε προτάσεις και για τους μηχανισμούς που μπορεί να υπάρξουν. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, περίπτωση που μας παρουσιάσατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, δεν ξέρω πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν σε αυτό το σχολείο, το οποίο πρόκειται τώρα να γκρεμιστεί. Δεν ε, είναι ζήτημα μόνο χρημάτων, είναι και ζήτημα ανθρώπων φυσικά. Είναι και ζήτημα βιολογικής ποικιλότητα Πράγματι τα βιοκαύσιμα είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα. Ο κύριος Πίμπαλξ ε, ήταν ε, κατά κάποιο τρόπο ιδρυτής, πατέρας όλων αυτών, αλλά ε, φαίνεται ότι θα πρέπει να υποστεί αυτό το ζήτημα σε περιορισμούς, τους οποίους δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε λοιπόν να αναθεωρηθεί το όλο ζήτημα. Δεν έχουμε χρόνο για να πω πολλά πράγματα. Θέλω και πάλι να τονίσω τη σπουδαιότητα του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια για αυτό. Εάν η ε, υπεύθυνη επιτροπή θέσει τα ζητήματα, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ, αλλά δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα δίκτυο βουλευτών, αλλά θα πρέπει να μένουν και πιστοί στις υποσχέσεις τους όταν ε, έρχονται και παρουσιάζουν στις επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Λόρο για την παρουσίαση. Κυρία Σνάιμπερ, επίσης ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Εδώ και πολύ καιρό ισχυρίζομαι ότι στο Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε έναν μόνιμο εισηγητή για τη συνοχή πολιτικής, κάποιον ο οποίος θα επιβλέπει τις διενέξεις και τη συνοχή ε, των έργων όλων των επιτροπών. Θα πρέπει να είναι ένας μόνιμος εισηγητής, ε, μια μικρή γενική διεύθυνση η οποία θα ε, δουλεύει αποκλειστικά για αυτό. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι να πάμε μπροστά. Ήθελα απλά να πω ότι χρειαζόμαστε επίσης συνοχή πολιτικής από τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς διότι αν παγώσουμε τους στόχους αμέσως ε, οι ενδιαφερόμενοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα έχουν αντίρρηση. Το ζήτημα δεν είναι τα βιοκαύσιμα ή μάλλον είναι το ζήτημα τα βιοκαύσιμα, αλλά και το πώς επιτυγχάνουμε τους στόχους, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να επιτύχουμε τους στόχους Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η δραστική, ε, ε, το δραστικό πάγωμα των στόχων θα δημιουργούσε πρόβλημα. Θα χρειαζόταν ε, κάποια συνεργασία, κάποια συνομιλία με τις ΜΚΑ ομικρών για την ενέργεια και με τους βουλευτές. Ε, κύριε Σνέντερ, Ιαστράμ, μπορείτε να... Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Ελπίζω ότι θα πέρασετε καλά στις διακοπές και θα επανέλθουμε σίγουρα μετά τις διακοπές για αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει πολλά να ξεκαθαριστούν ακόμη. Υπάρχει άλλωστε και το γραφείο αυτό ε, για επισήμανση ε, περιπτώσεων που υπάρχει έλλειψη της δέουσας συνοχής. Πριν το Δεκέμβριο θα υπάρξει δραστηριότητα πάνω σε αυτό. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε άλλες ερωτήσεις στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 29 Αυγούστου από τις 3 μετά έως τις 6 και μισή και μετά στις 30 Αυγούστου τις 9 έως τις 12.30. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ όλους και όλες